Ο Πρόεδρος, άρχεται η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί την 5η 18 Δεκεμβρίου 2008. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά 2009. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,